και κύριοι, παρακαλώ για την προσοχή σας. Ladies and gentlemen, your attention please. Παρακαλώ πάρτε τις θέσεις σας. Please take your seats. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. We're about to start. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει. Prime Minister Κυριάκος Μητσοτάκης has the floor. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. I would first of all like to thank uh... Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Φράου Μισελ, ο οποίο είχε την ιδέα να οργανώσει το ταξίδι αυτό, τον πρόεδρο τη Επιτροπή, Ούρσελα Φοντελάιν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντέβιτ Σασόλη, τον πρωθυπουργό τη ε, Κροατία, Ανδρέη Πλάνκοβιτ, που είναι μαζί, μου σήμερα, μαζί μας σήμερα εδώ, στον Εύρο, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αυτό που έχει συμβεί εδώ τις τελευταίες μέρες είναι επώδυνα προφανές σε όλους. Η Τουρκία κατά παράβαση τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία έχει ενθαρρύσει και έχει βοηθήσει δεκάδε χιλιάδε πρόσφυγε και μετανάστε να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Αλλά απέτυχε και θα συνεχίσει να αποτυγχάνει αν ακολουθήσει αυτή την στρατηγική. Δεν πρόκειται πλέον για ένα πρόβλημα προσφυγικό. Είναι μια κατάφορη απόπειρα από πλευρά Τουρκία να χρησιμοποιήσει απελπισμένου ανθρώπου να προωθήσει τη γεωπολιτική τη ατζέντα και να, ε, να στρέψει την προσοχή αλλού από την τρομερή κατάσταση στη Συρία. Οι δεκάδε χιλιάδε ανθρώπων που προσπαθούν που προσπάθησαν να εισέλθουν στην ε, Ελλάδα τις τελευταίε μέρες δεν ε, προέρχονται από την ΛΥΠ. Ζουν, εδώ και αρκετό καιρό με ασφάλεια στην ε, Τουρκία. Οι περισσότεροι μιλούν άπτεστα τουρκικά. Η Ευρώπη δεν θα υποκύψει σε εκβιασμού της Τουρκίας. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Τουρκία στην αντιμετώπιση του φυγικού προβλήματος και στην εξέβρεση μιας λύσης στο πρόβλημα της Συρίας, αλλά όχι από αυτές τις συνθήκες. Το καθήκον μου είναι να ε, υπερασπίσω την κυριαρχία της χώρας μου. Ταυτόχρονα η Ελλάδα ε, καλύπτει και εξυπηρετεί ιδιαίτερα και, της Ευρώπη, και την Ευρώπη, γιατί τα ε, σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και θα τα προστατέψουμε. Η ε, Ελλάδα αναμένει απτή αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ να σας πω ότι η παρουσία ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηγεσία εδώ στα ε, εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης θέλει ένα σαφές μήνυμα προς όλους. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Η Ευρώπη δεν έχει ανταπεξέλθει πλήρω στι υποχρεώσει για την ε, κάλυψη των αναγκών τη προσφυγική κλίση. Επίση, ότι αυτή η κρίση θα μα βοηθήσει όλου να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση καλύτερα με τους συναδέλφους μου είδαμε από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Μακριά από την ύπουλη προπαγάνδα των fake news που κυκλοφορούν για να κρύψουν την αλήθεια. Και αυτή είναι μία. Η Τουρκία κάνει πράξη την ομολογημένη απειλή της και επιχειρεί να στείλει δεκάδες χιλιάδες κατατρεγμένους ανθρώπους παρανόμως στην Ελλάδα ζητώντας ανταλλάγματα. Αν και ίδια έχει πλέον χαρακτηριστεί ασφαλής χώρα αποτελώντας de facto πλέον την πατρίδα πολλών από αυτούς, εξακολουθεί να τους χρησιμοποιεί ως γεωπολιτικούς μοχλούς για τους δικούς της σκοπούς. Παραβιάζει, παραβιάζει έτσι κατάφορα την κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την οποία οφείλει να συγκρατεί πρόσφυγες στο έδαφος της, αλλά και να εμποδίζει τις παράνομες οδούς προς την Ελλάδα. Δυστυχώς, η Τουρκία έχει μετατραπεί σε επίσημο διακινητή μεταναστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα δεν αποδέχονται αυτή την κατάσταση, την οποία αποδεικνύουν όλα τα τεκμήρια. δημόσιες δηλώσει του Προέδρου Ερντογάν με την απειλή ότι θα ανοίξει τις πύλες των μεταναστών προς την Ευρώπη. Τα βίντεο που δείχνουν δωρεάν μετακινήσει χιλιάδων ανθρώπων με τουρκικά λεωφορεία και συνοδεία στρατοφυλακή. Οι μαρτυρίες όσων έφτασαν στον Εύρο όπως και τα μηνύματα των δουλεμπόρων που γράφουν για δίθεν ανοιχτά σύνορα. Αγαπητοί φίλοι, το πρόβλημα αυτό δεν είναι πια προσφυγικό και μεταναστευτικό. Συνιστά μια ασύμετρη απειλή στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδος, που είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και η παράνομη εισβολή χιλιάδων ανθρώπων παίρνει τη μορφή της επιβολής του εθνικού μας εδάφους, με εμπροστοφυλακή συχνά ανθρώπους άγνωστης προέλευσης αλλά και αγνώστων σκοπών, που δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν απροκάλυπτα βία για να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια και εκτοξεύουν δακρυγόνα που χρησιμοποιεί ο τουρκικό στρατός. Είναι υποχρέωσή μου να περιφρουρήσω την ακαιρεότητα και την κυριαρχία της χώρας μου. Και αυτό θα κάνω. Ενώ είναι υποχρέωση της Ευρώπης να βοηθήσει την Ελλάδα και αυτό θα κάνει. Αντιδρούμε λοιπόν με γνώμονα την προστασία των συνόρων μας, αλλά και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Κινούμαστε απολύτως στο πλαίσιο του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Πάνω απ' όλα, ωστόσο, όσα συμβαίνουν στα ελληνικά σύνορα αποτελούν διεθνές πολιτικό ζήτημα πρώτου μεγέθους και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστούν. Από την πλευρά της η Ελλάδα έδειξε ότι μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της με όπλο την ομιμότητα και την αποφασιστικότητα. Μόνο στις τελευταίες μέρες οι δυνάμεις μας απέτρεψαν πάνω από 24.000 απόπειρες παράνομων εισόδων στον Εύρο και στο Αιγαίο. Προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις ανθρώπων που παραβίασαν τα σύνορα και πέτυχαν πολλές διασώσεις μεταναστών στη θάλασσα. Θέλω να συγχαρώ τις γυναίκες και τους άντρες της Ελλάς, των ενόπλων δυνάμεων, του λιμενικού για το έργο που επιτελούν αλλά και τους πολίτες που συμπαρίστανται αυθόρμητα στο δύσκολο έργο τους. Οι απειλές λοιπόν του κύριου Ερντογάν δεν πέρασαν. Προσέκρουσαν στην ενότητα του ελληνικού λαού. Στο φρόνημα και στην επιχειρησιακή ικανότητα των παιδιών του. Αλλά και στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Που είμαι σίγουρος ότι θα εκδηλωθεί ακόμα πιο αποφασιστικά τις επόμενες μέρες. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο προς όλους. Μην επιχειρείτε να μπείτε παράνομα στην Ελλάδα δεν θα τα καταφέρετε και αναλαμβάνετε ακέραια την ευθύνη των επιλογών σας. Η Ελλάδα έχει αποδείξει την ευαισθησία της, φιλοξενώντας πάνω από 100.000 ανθρώπους. Όμως ένα διεθνές πρόβλημα δεν μπορεί να το σηκώσει μόνο μια χώρα. Μάλιστα, όταν αργεί μια δίκαιη λύση, ο ανθρωπισμός μετατρέπεται σε αγανάκτηση. Γιατί η αλληλεγγύη δεν μπορεί να μένει μόνο στα λόγια. Άρα να απευθύνεται και προς τους Έλληνες πολίτες, των οποίων ήδη απειλείται η ασφάλεια, η περιουσία και η κοινωνική γαλήνη. Άλλωστε, βοήθεια στους κατατρεγμένους μπορεί να προσφέρει μόνο ένα κράτος. Δεν υπάρχει όμως κράτος χωρίς ασφαλή σύνορα. Και δεν υπάρχουν δικαιώματα χωρίς κράτους δικαίου. Η Ευρώπη μέχρι σήμερα απέτυχε να βρει κοινή λύση σε αυτό το σύνθετο πρόβλημα. Κάποιοι βολεύτηκαν να κλείσουν τα μάτια και να αφήσουν τα κράτη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα να αντιμετωπίσουν μόνα τους αυτή τη διαρκή κρίση. Η παρουσία σας εδώ είναι η καλύτερη απόδειξη ότι αυτό αλλάζει. Κλείνω ευχαριστώντας και πάλι τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη συμπαράστασή τους, η οποία σίγουρα θα γίνει και πιο έμπρακτη. Και τονίζω ξανά τη χαρά και την υπερηφάνεια την οποία ένιωσα δίπλα σε όσους υπηρετούν εδώ, στον ακριτικό Εύρο. Ήμουν, είμαι και θα είμαι κοντά τους, εκφράζοντας το σύνολο των Ελλήνων. Παραμένω όμως αισιόδοξο. Πρώτα η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι η Τουρκία μπορεί να βοηθήσει το προσφυγικό. Χρειάζεται τη στήριξη της Ευρώπης, όχι όμως υπό το κράτος απειλών. Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν εκβιάζεται, δεν εκβιάζονται, αντιδρούν και δεν προκαλούν, συζητούν. Και ελπίζω αυτό να συμβεί σύντομα σε κάθε περίπτωση όμως τα σύνορά μας είναι αδιαπραγμάτευτα, όπως αδιαπραγμάτευτη είναι και η θέλησή μας για μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα, οπλισμένη με το δίκαιο και τη λογική, θα πετύχουμε. Thank you again for your presence here. And let me now give the floor to the President of the Council, Charles Michel. Thank you. First of all, uh, dear Prime Minister, dear Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να επισκεφτώ τα ελληνικά σύνορα. Είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιε καταστάσει να μην μένουμε στι Βρυξέλλε, αλλά να βρισκόμαστε στο πεδίο και να έχουμε την καλύτερη δυνατή κατανόηση, να έχουμε την καλύτερη δυνατή αντίληψη του τι γίνεται και να, να δούμε τι γίνεται εδώ στα σύνορα με την Τουρκία. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω και επίση να εκφράσω την υποστήριξή μα στι ενέργειέ σα με τι δυνάμει ασφαλεία, με την ομάδα σας, με την κυβέρνησή σας τις τελευταίες αυτές τις ημέρες. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα και αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Είναι κρίσιμη σημασία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παρουσία μας εδώ μαζί στη χώρα σας σήμερα είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε στον ελληνικό λαό, στους Ευρωπαίους πολίτες και στον υπόλοιπο κόσμο ότι είμαστε μαζί, είμαστε μαζί γιατί θεωρούμε ότι η προστασία των συνόρων είναι ζωτική σημασία και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικά να ενεργούμε με αναλογικό τρόπο και να δείχνουμε σεβασμό στην ανθρώπινη ε, αξιοπρέπεια και στο διεθνές δίκαιο και εμπιστευόμαστε εσά, εμπιστευόμαστε την κυβέρνησή σα, γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και αν έχετε μπροστά σα ένα πάρα πολύ δύσκολο και πολύ πτυχικό ζήτημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό ω Ευρωπαίοι να προστατεύετε τα σύνορα μα και ταυτόχρονα όμω να επιδεικνύετε σεβασμό για το διεθνέ δίκαιο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, αναφερθήκατε σε πάρα πολλά σημαντικά θέματα και πράγματι έχουμε μία συμφωνία με την Τουρκία για το μεταστανευτικό. Και πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υλοποιείται αυτή η συμφωνία. Και γι' αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συνεχίσουμε να εγγυόμεθα την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και ε, θέλουμε και περιμένουμε από την τουρκική πλευρά να ε, σέβονται και να τηρούν αυτά που υποσχέθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένη συμφωνία. Αφορικά με τη Συρία, είναι σημαντικό να γίνουν όλες οι δυνατές προσπάθειες ώστε να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ευκαιρίες για μια πολιτική λύση, για μια διπλωματική λύση. Γι' αυτό επίσης υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες που γίνονται από τα ε, Ηνωμένα Έθνη έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες για να επιτύχουμε περισσότερη πρόοδος. Είναι μια τραγωδία, είναι μια πολύ μεγάλη τραγωδία για πολλούς ανθρώπους, οπότε ε, χρειάζεται η δέσμευσή μας για να δώσουμε περισσότερες ελπίδες και θετικές προοπτικές στο μέλλον. Ε, ο κ. Μπορέλ σήμερα βρίσκεται στην Άγκαρα για να περάσει το μήνυμα ε, το ευρωπαϊκό μήνυμα. Την Τετάρτη έχουμε μια συνάντηση στην, στις Βρυξέλλες με τους, ε, ευρωπαϊκού, με τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εσωτερικών και στην Παρασκευή έχουμε συνάντηση στην Κροατία με τους Υπουργού Εξωτερικών. Αυτό σημαίνει ότι δρούμε, ενεργούμε, είμαστε ε, μαζί, είμαστε ενεργοί και στις επόμενες ημέρες, στις επόμενες εβδομάδες θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με εσά, με τη δική σας κυβέρνηση, με όλους τους ευρωπαϊκούς φορούς, ώστε να δείξουμε ότι είμαστε σε θέση να προστατεύουμε τα σύνορά μας, ότι είμαστε είμαστε σε θέση να δείχνουμε την ενότητα όταν πρέπει να είμαστε ισχυροί, δυνατοί και μπορούμε να είμαστε σε θέση να δείχνουμε ότι αυτό είναι εφικτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυριακό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πράγματι, ε, ζούμε εξαιρετικές ε, καταστάσεις και μόλις επισκεφτήκαμε τα σύνορα και είδαμε πόσο έντονη και δύσκολη είναι η κατάσταση. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πάρα πολύ δύσκολη ε, αποστολή στην συγκράτηση της κατάστασης αυτής και την αντιμετώπιση της κατάστασης και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Έλληνες συνοριοφύλακες και το λιμενικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολίτες, ε, τους ε, αστυνόμους και τη Frontex για τις άοκνες προσπάθειές τους. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και να σας πω ότι οι ελληνικές ανησυχίες είναι δικές μας ανησυχίες. Τα σύνορα αυτά δεν είναι μόνο ελληνικά ε, σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και βρίσκομαι εδώ σήμερα ως Ευρωπαία στο πλευρό σας. Θέλω επίσης να ε, εκφράσω τη συμπόνια μου για τους μετανάστες οι οποίοι ε, πέσαν στην παγίδα των ψεύτικων υποσχέσεων και βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να δώσουν, στείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα. Να δηλώσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και υποστήριξη προς την Ελλάδα η πρώτη προτεραιότητα είναι να φροντίσουμε ότι θα τηρηθεί τάξη στα ελληνικά εξωτερικά σύνορα, που είναι και τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρώπη. Ε, είμαστε δεσμευμένοι να κινητοποιήσουμε όλη την απαραίτητη επιχειρησιακή υποστήριξη στι ελληνικέ αρχέ. Κατόπιν ε, αιτήματο ε, τη Ελλάδο, η Frontex ετοιμάζεται να αναπτύξει μια ομάδα παρέμβασης, παρέμβαση. παρέμβασης θα αναπτυχθεί θα αναπτυχθούν 7 σκάφη, 2 ε, ελικόπτερα, 1 αεροσκάφος, 2 ε, οχήματα με κάμερες, 100 συνοριοφύλακες, πλέον των ε, ήδη υπάρχουν 530. Οι συνοριοφύλακες θα αναπτυχθούν από τη Frontex στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Δεύτερον, μπορούμε να παρέχουμε οικονομική υποστήριξη 700 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα ε, είναι 350 εκατομμύρια ευρώ που είναι διαθέσιμα άμεσα και επιπλέον 350 εκατομμύρια ε, ευρώ τα οποία μπορούν να ζητηθούν ε, στο πλαίσιο ενός τροποποιητικού προπολογισμού. αυτό, αυτή η υποστήριξη αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού και για τη δημιουργία του απαραίτητου ε, Τη απαραίτητη υποδομή. Ξεκινάμε τον μηχανισμό πολιτικής προστασία βάσει αιτήματο που έχει υποβληθεί από την Ελλάδα. Μέσω αυτού του μηχανισμού η Ελλάδα μπορεί να λάβει βοήθεια αναφορικά με ιατρικές ομάδες, ιατρικό εξοπλισμό, ε, σκηνές, ε, κουβέρτες, ό,τι χρειάζεται. Κυριακό, Σάρλ, Νταβίδε, Αντρέ και εγώ θα ε, είμαστε σε πολύ στενή επικοινωνία τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες για να διασφαλίσουμε ότι θα προσφέρουμε κάθε απαραίτητη υποστήριξη. Η κατάσταση στα σύνορά μας δεν είναι μόνο ένα θέμα το οποίο πρέπει να χειριστεί η Ελλάδα μόνη της, είναι ευθύνη της Ευρώπης συνολικά και θα διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα με, με τάξη, ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα. Όσοι προσπαθούν να δοκιμάσουν την ενότητα της Ευρώπης θα απογοητευθούν. Θα διατηρήσουμε τη γραμμή μας και η ενότητά μας θα κυριαρχήσει. Τώρα χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες και ψύχρεμες δράσεις και ε, δράσεις με βάση τις αξίες μας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός και οι άνθρωποι δεν αποτελούν μόνο ε, αυτό σκοπό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε στις επόμενες ημέρες. Εγώ ευχαριστώ την Ελλάδα που είναι η δική μας ευρωπαϊκή ασπίδα σε αυτούς τους καιρούς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, τους συναδέλφους. Είναι πολύ σημαντικό το ότι βρισκόμεθα σήμερα εδώ μαζί πολιτική εκπροσώπηση, ε, κοινοβούλιο, ευρωκοινοβούλιο, ελληνική κυβέρνηση. Αν θέλαμε να επιστρέψουμε στις Βρυξέλλες και τα πράγματα συνεχίζονταν όπως εξακολουθητικά έγιναν μέχρι σήμερα, πιθανότατα και αυτό θα καθίστατο μία ανώφελη ευκαιρία, διότι εμείς έχουμε ανάγκη ενός πράγματος και το βλέπουμε καθημερινά να ενισχύσουμε μια κοινή πολιτική για το μεταναστευτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πραγματικά είμαι πάρα πάρα πολύ ανήσυχος ότι πολλοί κυβερνήσεις να μην συναισθάνονται, να μην συνειδητοποιούν πριν από 1,5 χρόνο αν είχαμε ακούσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαμε ακολουθήσει την ε, μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, πιθανότατα σήμερα, δεν θα αντιμετωπίζαμε αυτές τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Για το Ευρωκοινοβούλιο που έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται στην Ευρώπη, δεν έρχεται μόνο το να πάει στην Ιταλία, στη Μάλτα ή στην Ισπανία έρχεται στην Ευρώπη και οφείλει να είναι η Ευρώπη η οποία θα πρέπει να ασκήσει μεταναστευτική πολιτική, να συμμεριστεί το βάρος του μεταναστευτικού, να ανακατανείμει ισοδύναμα που θα εγγυάται το γεγονός ότι στην Ευρώπη είναι εγγυημένε οι ελευθερίες και τα δικαιώματα των ατόμων. Αν όμως δεν έχουμε μια κοινή πολιτική στο μεταναστευτικό, πώς θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε όλα τα όσα ανέφερα και να είμεθα και υπερήφανοι επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε μια καμπή και η σημερινή παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής, του Συμβουλίου και η παρουσία του Ευρωκοινοβουλίου τούτο θέλουν να πούν ένα κάλεσμα στην Ευρώπη να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα την πιθανότητα να υπάρξει κοινή πολιτική στο μεταναστευτικό. Συγχρόνως βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να πούμε ευχαριστώ στην Ελλάδα, στους Έλληνες πολίτες, σε όλους όσοι προσπάθησαν και προσπαθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό και όχι σήμερα να προστατεύσουν ανθρώπους, να μην σορεύονται δεινά και βάσανα. Αλλά βρισκόμαστε σήμερα εδώ και για ένα τρίτο λόγο να πούμε στην Τουρκία ότι εμείς θέλουμε να συνδιαλλαγούμε, να συζητήσουμε και ότι θα πρέπει να σεβαστεί τις συμφωνίες. Πιστεύω ότι αυτό είναι το σημάδι για το Ευρωκοινοβούλιο αυτής της επίσκεψης, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στις Βρυξέλλες και αυτή είναι η δέσμευση που οφείλουμε να αναλάβουμε για να σχηματίσουμε, να χαράξουμε μια κοινή πολιτική. Αυτό είναι που μας ζητούν οι Έλληνες πολίτες σήμερα, οι μεσογειακοί λαοί και όλοι οι λαοί της Ευρώπης σήμερα να αντιμετωπίσουμε μια πρόκληση που δεν θα αναλωθεί σε ένα χρονικό γράφημα, αλλά να καταστεί μέσω μακροπρόθεσμη στρατηγική. Επιτρέψτε μου τώρα μια σκέψη, διότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάμπολοι χιλιάδες ανηλίκων, ανήλικα ασυνόδευτα και εγώ νομίζω ότι μια δέσμευτη που οφείλω να αναλάβω και ομού μαζί με τους άλλους θεσμούς είναι να έχουμε μια στρατηγή για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, τα συνόδευτα ανήλικα. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε το μέλλον τους, να προστατεύσουμε το μέλλον τους και πιστεύω ότι επ' αυτού η δέσμευση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων οφείλει να είναι πολύ εντονότερη εξ όσων υπήρξε σήμερα λόγω γενιοδορίας, διότι πολύ συχνά οι πολιτικές ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων υπήρξαν πραγματικά δεν βασίστηκαν στη γενοδορία, αλλά στο δικό του συμφέρον. Πιστεύω ότι ο ευρωπαϊκό χώρο αξίζει κάτι περισσότερο και πιστεύω ότι αυτό είναι ο τρόπο για να σεβαστούμε τη μεγάλη δέσμευτη που οι αρχέ, οι θεσμοί και οι Έλληνε ε, κάτοικοι υλοποιούν αυτή τη στιγμή. Σα ευχαριστώ για την, για την προσοχή σα. Ευχαριστώ κύριε Πρωτάνδρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κυριάκο. Κυρίες και κύριοι, Ούρσουλα Σάρλ Κάρλ Ντάβιντεφ, εκ μέρους της ε, Κρατικής Προεδρίας του Συμβουλίου, ε, ήρθαμε σήμερα εδώ πρώτον για να εκφράσουμε την ε, αλληλεγγύη μας και την υποστήριξή μας στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά να να επίση την κοινή ευρωπαϊκή αποφασιστικότητά μα να βοηθήσουμε την Ελλάδα και να βρούμε μια ευρωπαϊκή ε, απάντηση σε αυτή τη, τη νέα μεταναστευτική, τη νέα, νέα κατάσταση και ελπίζουμε δεν θα εξελιχθεί σε κρίση. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κυριάκο που άλλαξε την πολιτική της Ελλάδας στην προστασία των, σημερα, των σύνορων, δηλαδή να μην επιτρέπει την παράνομη μετανάστευση στην επικράτητά της, γιατί όπως είπε η Ούρσουλα η Ελλάδα είναι η ασπίδα, τα πραγματικά εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και ο εγγυητής της σταθερότητας για την, Ευρω... για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το λέω αυτό και ως Πρωθυπουργό, ο οποίος μιας χώρας που ε, βρίσκεται στη, στη, διαδρομή τη, τη, τη, των Δυτικών Βαλκανίων. Οπότε είναι προσόφερος όλων μας τα ελληνικά ε, σύνορα να μην είναι ποροδί και συνεπώς εκτιμούμε πάρα πολύ και την ενημέρωση της προσπάθειας ε, της ελληνικής αστυνομίας και των ανδρών και γυναικών, των δυνάμεων ασφαλείας και του στρατού. Είναι μαζί μου ο Υπουργό ε, Εσωτερικών, ο οποίος θα είναι, θα είναι πρόεδρος της ε, έκτακτης έλευση του Υπουργών Εσωτερικών. Είναι ένα σήμα ότι ενεργούμε έγκαιρα και στέλνουμε τα σωστά μηνύματα, μηνύματα υποστήριξης, ακόμα και με τις ομάδες ταχεία παρέμβαση που μπορούν να αναπτυχθούν με την συνεισφορά της ε, Frontex και της EASO, καθώς επίσης και την οικονομική ε, βοήθεια που ε, είπε, όπως είπε η Ρούσιλα είναι ήδη διαθέσιμη. Ε, ταυτόχρονα στέλνουμε ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι οι καλές σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζονται και στις ενέργειες και των δύο μας. Θα αναζητήσουμε μια πολιτική και διπλωματική λύση η οποία θα αποκλιμακώσει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα εδώ στις Καστανιές ε, και την κατάσταση που είδαμε πριν από μερικές ώρες. Ε, η υποστήριξή μας ως Προεδρίας θα είναι να είμαστε αποφασισμένοι, δεσμευμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και να ε, αποτρέψουμε την επανάληψη του 2015-2016. Έχω πει πολλές φορές ότι κανένα άλλο φαινόμενο δεν έχει επηρεάσει το πολιτικό τοπίο της Ευρώπης και των κρατών μελών της, όπως η μεταναστευτική κρίση την οποία είδαμε τα τελευταία 4 ή 5 χρόνια. Συνεπώ, θα πρέπει να πάρουμε τα μαθήματα από το παρελθόν και από την εμπειρία αυτή, να μείνουμε μαζί, να κρατήσουμε τη γραμμή μα και να υποστηρίξουμε τι προσπάθειε τη ελληνική κυβέρνηση, τι οποίε ε, είδαμε δύο όμαση. Ευχαριστώ, Αντρέη. Ε, θα ήθελα να κλείνω να σας ευχαριστήσω όλου που βρίσκεστε εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την έκφραση τη αλληλεγγύη από όλου του θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Ελλάδα, προ τον ελληνικό λαό, τι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει, την ελληνική αστυνομία για τη δουλειά που κάνουν στην προστασία των ε, συνόρων τη Ευρώπη. Όπω είπε, Αντρέ, η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί μια διαφορετική διαδρομή σε ό,τι αφορά την προστασία των συνόρων. Και στέλνουμε ένα πάρα πολύ σαφέ μήνυμα ότι οι μετανάστε και οι πρόσφυγε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω πιόνια, ω όργανα σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι είναι τα πραγματικά θύματα τέτοιων πολιτικών και αυτή είναι μια ε, προσέγγιση η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή. Αν η Ευρώπη θέλει να προστατεύσει του πολίτε, πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει τα σύνορά μα. Και αυτό που εμεί με την Ιταλία, με την Ισπανία, με άλλε χώρε που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουμε. Ταυτόχρονα όμω δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μα. Ο όλος σκοπός, όλος στόχος της ε, δημιουργίας της Frontex είναι για να μοιραστούμε το βάρος της προστασίας των συνόρων και, και, και κάθε βοήθεια που μπορεί να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, ευπρόσδεκτη γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Ταυτόχρονα το γεγονό ότι είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα σύνορα μα και να περιορίσουμε την παράνομη μετανάστευση στο μέγιστο βαθμό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να, να, να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό σε ό,τι αφορά την αλλαγή των ε, υφιστάμενων πολιτικών ασύλου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας ε, ενοχλεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να είμαι λίγο προκλητικός και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει σοφά το χρόνο που πέρασε από την τελευταία μεταναστευτική κρίση για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κατάσταση. Ήρθε ο καιρό όμω να το κάνουμε. Πρέπει να είμαστε σε θέση να δείξουμε αποτελεσματικά ότι μοιραζόμαστε το βάρο, στην αντιμετώπιση του προβλήματο. Χρειαζόμαστε διάφορου τύπου τύπους ε, πολιτικών. Πρέπει να σκεφτούμε πρωτότυπα και καινοτόμα. Και για να είμαι ειλικρινή, δεν μπορούμε ε, να έχουμε τόσες χώρες ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε περνάνε και σπρώχνουν το βάρο τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων σε αυτέ τι χώρε που από γεωγραφία και μόνο βρίσκονται στη θέση που βρίσκονται ενώ ταυτόχρονα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προβλήματος αυτό ιστορικά και ξέρω ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες ιδέες που προετοιμάζει η Επιτροπή ε, και θέλουμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε στο να επιτευχθεί μία λύση σε αυτό το πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω όλους που βρίσκεστε εδώ σήμερα είναι ε, δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας. Ε, πολλοί άνθρωποι ε, εξάγρυπνοι τις τελευταίες τρεις-τέσσερις ημέρες για να κάνουν τη δουλειά τους, να την κάνουν σωστά. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, μπορούμε να προστατεύσουμε τα σύνορα, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα σύνορα και ειλικρινά ελπίζω τώρα, ότι τώρα που η απειλή της αποστολής εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στην Ευρώπη έχει υλοποιηθεί, αλλά αν επιτυχώς ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε μια νέα προσέγγιση. Ε, είναι το λιγότερο που οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που πολλές φορές νιώθουν ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν και σήμερα χρησιμοποιούνται ως όργανα, ως πιόνα για την προώθηση άλλων φιλοδοξιών. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Σας εδώ σημαίνει πάρα πολλά στην κυβέρνηση, αλλά κυρίως σημαίνει πάρα πολλά στο λαό, στους ανθρώπους που ζουν εδώ, σε αυτή τη γωνιά της Ελλάδας, στον Εύρο. Σημαίνει πολλά σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ.